Yeah, just while, just while we're sitting here and waiting for... Um, Καθώς περιμένουμε, λέει η πρόεδρος Μακάβαν, την επιτροπή που κάπου κόλλησε στην κυκλοφορία, θα έρθει όμως με τα πόδια. 18 και 45 συνέρχεται η DEG, Democracy Support Group για τη Ζιμπάμπουε και με, ε, ζήτημα, με θέμα μάλλον παρατήρηση εκλογών. 18 και 45, δεν θυμούμε ακριβώς πού, αν κάποιος ξέρει, μπορούμε να σας πούμε. Μαριέτα. A3G2 Στην αίθουσα Α3G2, G2, αν θέλετε να έρθετε να ακούσετε και να μιλήσετε για τη Ζιμπάμπουε. Τώρα, αγαπητές και αγαπητοί, ας πάμε στο 22 στην ε, ημερήσια διάταξη της ε, Επιτροπής ε, Αναπτύξεως και εκεί προβλέπεται κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εδώ θα συνδιευθύνω τη συζήτηση με τον συνάδελφό μου, κύριο Αχτουι, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Παρόντες είναι και συνάδελφοι συνεισηγητές για την ε, νομοθέτηση για το ε, σχέδιο, σχεδιασμό εξωτερικών επενδύσεων. Θα συζητήσουμε σήμερα την πρόοδο του σχεδίου εξωτερικών επενδύσεων, νομοθέτημα το οποίο ε, συμφωνήθηκε μεταξύ τριών κοινοβουλευτικών επιτροπών και νομίζω μάλιστα ότι ήταν μια χαρά η συνεργασία αυτή και θέλουμε τώρα να δούμε πόσο καλά εφαρμόζεται η νομοθεσία αυτή. Να δώσω το λόγο αμέσως στον πρόεδρο Ατουή για να σας απευθύνει τον χαιρετισμό της Επιτροπής Προπολογισμών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητές και αγαπητοί Πρόεδροι, πράγματι το 2017 οι ε, επιτροπές, οι τρεις επιτροπές προϋπολογισμών εξωτερικών και αναπτύξεως συνεργάστηκαν και οι τρεις συνεισηγητές ε, έκαναν ε, μια σπουδαία δουλειά, την οποία στηρίξαμε, διότι θεωρούμε ότι είναι μια συνολική ανταπόκριση αυτού του μηχανισμού που θα μας επιτρέψει ίσως να αρχίσουμε να συμβάλλουμε σε μια λύση του μεταναστευτικού προβλήματος του μεταναστευτικού προβλήματος που ακόμα στο μεγαλύτερο μέρος του το έχουμε μπροστά μας και που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη με πολύ θάρρος. Ο μηχανισμός αυτός ε, ανταποκρίνεται στις ε, προσδοκίες μας. Ποιες είναι οι πρώτες εφαρμογές, εντάσσεται σε μια ευρύτερη και καλύτερη στρατηγική και συνεργασία μεταξύ των διαφόρων άλλων μέσων και μηχανισμών, με συμμετοχή νέων φορέων και πραγματικά συμβάλλει σε αυτή τη μόχλευση, μόχλευση άλλωστε και για ένα πιο εμβαθυμένο πολιτικό διάλογο. Και Άλλο ερώτημα, ε, προσφέρουμε την αναγκαία ε, διοικητική υποστήριξη στους εταίρους μας και ιδίω στην Αφρικανική Ήπειρο. Ιδού λοιπόν κάποια πρώτα στοιχεία, κάποια πρώτα ερωτήματα ε, στα οποία θα θέλαμε να ακούσουμε απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που επιτρέπετε να συμμετάσχουμε στην κοινή αυτή συνεδρίαση των Επιτροπών μας. Η Πρόεδρος Μακάβα. Υπενθυμίζω στου και στι συναδέλφους ότι όταν διαπραγματευθήκαμε το σχετικό νομοθέτημα επέμεινε το Κοινοβουλίο στο γεγονό ότι δεν πρόκειται για άλλο ένα ε, ταμείο ε, δανειοδοτήσεων αλλά έχει ως στόχο την μείωση της φτώχειας που είναι στόχος της ανάπτυξης και θέλουμε να φτάσουμε σε μέρη όπου δεν φτάνουν άλλα ε, δανειοδοτικά ταμεία και γι' αυτό μιλούμε και για εγγύησεις χωρίς να απολογώ να δώσω το μικρόφωνο στην Μαριέτα Γιάγκερ που για δεύτερη φορά έρχεται σήμερα στην ε, συνεδρίαση της Επιτροπής μας και την ευχαριστώ πολύ για την έξτρα αυτή προσπάθεια που καταβάλει. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητή Λίντα, αξιότιμες και αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Ε, χαρά μου που βρίσκομαι εδώ για δεύτερη φορά και βέβαια η Επιτροπή είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή, που μπορεί να συζητήσει μαζί σας για την εφαρμογή του External Investment Plan, η IP, το οποίο διαπραγματευτήκαμε μαζί με τις τρεις προαναφερθήσεις κοινοβουλευτικές επιτροπές και μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να είναι ευγνώμων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συνεργασία αυτή. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν. Η διαπραγματεύσεις υπήρξαν επιτυχείς. Ο κανονισμός άρχισε να ισχύει από τον Σεπτέμβριο. Ήσασταν παρούσα και στο Strategic Board Meeting και έκτοτε έχουμε δημοσιεύσει δύο προσκλήσεις εκδηλώσεων ενδιαφέροντος. Ε, μία τέλη Ιανουαρίου για δύο παράθυρα των εισαγωγικών για τη βιώσιμη ενέργεια και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δεύτερη ε, πρόσκληση εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για άλλα ε, παράθυρα για τη γεωργία, την ψηφιακή οικονομία και τα αστικά κέντρα. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση μπορώ να σας ενημερώσω ότι το, εξωτερικό, μάλλον σχέδιο εξωτερικών επενδύσεων αποτελεί μεγάλη επιτυχία. Κυρία Πρόεδρε, 12 συνολικά φορείς εταίροι έχουν προτείνει προγράμματα επενδύσεων στα πέντε αυτά, στις πέντε αυτές θηρίδες επενδύσεων που σας ανέφερα προηγουμένως. 46 συνολικά προτάσεις έχουμε λάβει και αναμένονται άλλες δύο συνολικά αξίες 3,5 δισεκατομμύριων για πέντε θηρίδες. Θα θυμάστε κυρίες και κύριοι ότι η εγγύηση που έχουμε είναι για 1,5 δισεκατομμύριο. Αυτό σημαίνει ότι οι προσδοκίες και προτάσεις των εταίρων μας είναι σχεδόν διπλάσεις από αυτό που διαθέτουμε, από το ποσό εγγύησης που διαθέτουμε. Τα 2,5 δισεκατομμυρία και ε, κινούνται προς την κατεύθυνση του, ε, ε, του παραθύρου για τα ψηφιακά και 16 bips για τα άλλα. Και αιτήσει για ένα δισεκατομμύριο έχουμε λάβει για τις άλλες τρεις θηρίδες, πέντε για τη γεωργία, αστικά κέντρα έξι και ψηφιοποίηση τέσσερα Επί του παρόντος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί τις προτάσεις, η δε επιλογή βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια που ε, καθορίσαμε όλοι μαζί στον κανονισμό. Οι πρώτες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένονται για Μάιο-Ιούνιο αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα αρχίσουμε την, με, συνάντηση τεχνικής αξιολόγησης την Παρασκευή 27, δηλαδή μεθαύριο, για τις ε, δύο πρώτες θηρίδες και μετά από συζητήσεις με τις χώρες μέλη και το ε, Επιχειρησιακό Συμβούλιο ε, θα επανέλθουμε στις 20 Ιουνίου για την συνάντηση του Στρατηγικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Στρατηγικής μάλλον. Και θα προχωρήσουμε μετά το με, στην πλήρη εφαρμογή για το 2018. Δηλαδή, για να εκπληρώσουμε πλήρως τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό. Βέβαια, μπορώ να συνεχίσω επάπειρον στην ουσία. Βλέπω ότι μόλις ήρθε η Καταρίνα Μαρτένοβα από την Αρμόδια Γενική Διεύθυνση. Θα ήθελα ωστόσο να σας διαβεβαιώσω ότι για να ελοποιήσουμε τα προβλεπόμενα από τα EIP συνεργαζόμαστε με τις αντιπροσωπείες μας, διότι επιμένουμε ότι πρόκειται για κοινό εγχείρημα και θέλουμε βέβαια διαθρωμένο και διαρκή διάλογο, όχι μόνο με τους τοπικούς παράγοντες, αλλά και με τις ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες στις ε, χώρες εταίρους, για να ενισχύσουμε και τις ιδιωτικές επενδύσεις και να βελτιώσουμε το επενδυτικό κλίμα. Επισημαίνω επίσης ότι βλέποντας τον μεγάλο αριθμό ετοιμάτων για ΠΙΠ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξέτεινε την πρόσκληση και προς τις χώρες να συμμετάσχουν και να ε, προσφέρουν και άλλα κονδύλια για εγγύησεις. Έχουμε πρόσθετες λοιπόν συμβολές από Εστονία, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία και βέβαια και από το Ίδρυμα ε, του Ζεύους Γκέιτς. Έχουμε και άλλους λοιπόν εταίρους οι οποίοι συμμετέχουν στον ε, σχεδιασμό και εξασφαλίζοντας έτσι την ε, επιτυχή έκβαση των προσπαθειών του. Από σας θα εξαρτηθεί κυρία Πρόεδρε αν θέλετε να ε, συνεχίσω αλλιώ να λάβει τώρα τη σκητάλη συναδελφός μου της DG Near διότι βέβαια συνεργαζόμαστε και μοιραζόμαστε τις προσπάθειες. Και εξέρω τη συνεργασία όλων των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άλλωστε, συνεργαζόμαστε για τον δεύτερο και τρίτο πυλώνα του EIP, δηλαδή κάνουμε καταγραφή της τεχνικής βοήθειας και προωθούμε πολιτικό διάλογο για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι έχουμε στην εργαλειοθήκη μας ώστε το, ο ευρωπαϊκός ε, επενδυτικός σχεδιασμός να ε, αποβεί επιτυχής. Σας ευχαριστώ. Εσείς επιθυμείτε να λάβετε το λόγο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως μόλις εξήγησε η Μαριέτα, δεν πρόκειται μόνο για ένα κοινό εγχείρημα, είναι και εγχείρημα το οποίο έχει και τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βλέπω εδώ και τους βασικούς συνεισηγητές οι οποίοι έχουν βοηθήσει να μεγαλώσει το μικρό αυτό παιδάκι. Η περίοδος εφαρμογής δεν έχει αρχίσει ακόμη, αλλά ο ρυθμός ανταπόκρισης και η προθυμία των άλλων φορέων να συνεργαστούν μαζί μας αποτελούν δείγμα ε, ταχύτητα της πρόοδου. Κάποιες προτάσεις είναι ισχυρότερες ας πούμε από άλλες αλλά έχουμε σημαντικό στοιχείο καινοτομία. Ορισμένες προτάσεις ε, κατευθύνονται ιδίω σε μεταναστευτικούς πληθυσμούς, ε, άλλες για τις διάφορες διασπορές και αναμένουμε με ενδιαφέρον την πρώτη τεχνική συζήτηση που θα διεξαχθεί για τις δύο πρώτες ε, θηρίδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ενεργειακή αποδοτικότητα και διασυνδεσιμότητα. Αυτά θα γίνουν θα συζητηθούν την Παρασκευή που μας έρχεται και αργότερα τον Μάιο τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπε θεωρούμε ότι υπάρχει ήδη μια καλή βάση για να γίνει και πρόοδος επιτόπου. Η εγγύηση είναι ο τομέας όπου διδασκόμαστε καθώς προχωρούμε από τις προσπαθίες μας. Έχουμε ωστόσο όλα τα στοιχεία, όλα τα συστατικά αν θέλετε, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι επιτυχές για το μέλλον. Για το ίδιο το blending, το μείγμα, από την πλευρά τη δική μας Digineer, είναι ένας καλολαδωμένος μηχανισμός, έχουμε συμμετοχή όλων των εταίρων στους οποίους στραφήκαμε και προάγουμε και την καινοτομία εν προκειμένου στηρίζουμε και policy operations και investment operations και όπως είπε και η Μαριέτα διεξάγουμε διάλογο πολιτικής με τις χώρες εταίρους και για το επενδυτικό κλίμα, για ζητήματα επενδυτικού κλίματος δηλαδή, αλλά και για ευρύτερες ανάγκες περιβάλλοντος πολιτικής ας πούμε. Θα σταματήσω εδώ και είμαι στη διάθεσή σας. Πρόεδρος Μακάβαν, για τι είδους έργα μιλούμε και πού. Ωστόσο ας λάβουν πρώτα το λόγο οι Μήπως έχετε πρώτα ερωτήσεις. Εσείς κύριε Κούκαν. Thank you very much for the information. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις. Η πρώτη, όπως έλεγε σωστά Πρόεδρε, μπορούμε να έχουμε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για το τι είδους έργα υποβάλλονται. Άλλη ερώτηση που εν μέρη απαντήθηκε είναι ότι ορισμένα κράτη-μέλη είναι έτοιμα να συμβάλλουν αλλά πόσα επιπλέον χρήματα έβαλαν σε αυτήν την εγγύηση για να μπορέσουν να εγγύθουν αυτά τα έργα. Και επίσης θα ήθελα να γνωρίζω όταν θα ορίσουμε τις επενδυτικές ευκαιρίες, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα ισχύουν όλα τα κριτήρια, ας πούμε κλιματικές αλλαγές 28%, ειδική προσοχή στις χώρες που είναι λιγότερο αναπτυγμένες. Επίσης, έχουμε συμφωνήσει σε κανόνες για τις μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες, δηλαδή σχέσεις με αυτές τις χώρες, να δούμε πώς προχωρούν ε, στην θέσπιση αυτών των δυνατοτήτων των επενδυτικών. Και έπειτα για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και περιμένουμε την πρόταση της Κομισιόν ακούγονται, ακούγονται διάφορες φήμες δεξιά και αριστερά αλλά ακούσαμε και κάποιες πιο βάσιμες φήμες ότι θα υπάρχει ένα μέσο, ενιαίο μέσο εξωτερικών επενδύσεων που θα καταπιεί ε, και θα συνδυάσει διάφορα κονδύλια που υπάρχουν τώρα. Πώς θα γίνει λοιπόν όλο αυτό όσον αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη. Κύριος Φρουντζουλίκα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εξ όσων γνωρίζω, κανονικά η ΕΤΕΠ θα πρέπει να δώσει γραπτή γνωμοδότηση για τα θέματα αυτά που θα συνοδεύει κάθε πρόταση επενδυτικού παράθυρου. Ερώτησή μου είναι αν η Κομισιόν έχει λάβει αυτές τις, ε, προ, γραπτές και αν είναι δημοσιευμένες και αν μπορούμε να τις έχουμε. Δεύτερον, αναφέρατε ότι λάβαμε πολλές προτάσεις κτλ. κτλ. Εσείς είστε σίγουροι, δηλαδή η Κομισιόν να είναι σίγουροι ότι ένα σημαντικό κομμάτι αυτών των πόρων θα χρησιμοποιηθεί από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Πρόεδρος, να προσθέσω κι εγώ μια ερώτηση που ίσως θα έπρεπε να την είχα θυμηθεί, αλλά όταν φτιάξαμε την νομοθεσία, αν τα κάτι μέλη συμβάλλουν στο Ταμείο, έχουν επιπλέον δικαιώματα και τι γίνεται με το Ίδρυμα, με το Ίδρυμα Bill Gates που κάνει κάποια δωρεά. Τι σημαίνει αυτό, μπορείτε να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει σε αυτό το πλαίσιο. Άλλες ερωτήσεις. Όχι. Μαρία, τα παρακαλώ. Ευχαριστώ, Λίντα. Μπορώ να σας δείξω τον κατάλογο των έργων αν θέλετε, μπορώ να σας δείξω και τις υποβολές, αλλά πιθανότατα ε, δεν έχουμε αρκετό χρόνο να το κάνουμε αυτό τώρα. Όπως είπε η Κατερίνα, υπάρχουν πολλές ε, καινοτόμες προτάσεις, όπως αυτή που αφορά την διασπορά που βλέπουμε μεγάλο δυναμικό όταν βλέπουμε την, τα έτη της μετανάστευσης όπου η διασπορά βασικά συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στη χώρα προέλευσης. Επίσης βλέπουμε νέα project όπως το Room to Run που, προτείνει την ασφάλιση ε, των ιδιωτικών ε, επενδύσεων αλλά και νέες προτάσεις ε, για την Αφρική με την Ζάμπια σε πιλωτικό πρόγραμμα πούμε, για, τη για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έχουμε ένα πρόγραμμα επίσης για τη γειτονία πρέπει να εξασφαλίσουμε και γεωγραφική ισορροπία όπως είπαμε αλλά βεβαίως εξασφαλίζουμε ότι όλα τα κριτήρια του κανονισμού θα τηρηθούν όχι μόνο 28% για τις κλιματικές αλλαγές, όχι μόνο για την μετανάστευση, ισότητα των φύλων και θα εξασφαλίσουμε ότι συμβάλλουμε για την τήρηση όλων των προτεραιοτήτων. Και βασικά ο κύριος στόχος, δηλαδή να χρηματοδοτηθούν λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και τα ευάλωτα περιβάλλοντα. Ε, πώς θα το κάνουμε αυτό, ε, εστιάζουμε την παροχή, τις διατάξεις μάλλον το, της Συμφωνίας Περιεγγύσεων, δεν μπορώ να σας πω τώρα όλες τις λεπτομέρειες, αλλά μπορώ να σας πω ότι λέει ας πούμε 30% πρέπει να πάνε στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρε. 20% ευάλωτες χώρες. Έχουμε βάλει κάποιες προϋποθέσεις στη Συμφωνία Περιγγύσεων ότι θα σας εξασφαλίσουμε και όλους τους φορείς ώστε να τηρηθούν τα κριτήρια και οι στόχοι του κανονισμού. Αυτή είναι η πρόθεση για το πώς θα εξασφαλίσουμε την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού και των κριτηρίων του. Συν τις πολιτικές υποχρεώσεις που αναλάβαμε. Τώρα, όσον αφορά τις συμβολές, ναι, βεβαίως θέλαμε περισσότερα κράτη-μέλη να συμβάλλουν. Α, ναι, πόσα χρήματα, ναι. Ε, ε, ε αυτό ήθελα να το, να το κρατήσω μυστικό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι μια συμβολική συμβολή, αλλά είναι μια αρχή. Μιλάμε για 100.000 από την Εστονία, 300.000 από την Τσεχία, 1 εκατομμύριο από τη Γερμανία και από το Ίδρυμα Bill και Melinda Gates ανακοίνωσαν τη συμβολή 50 εκατομμυρίων δολαρίων που μας κάνει σε ευρώ 42,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά έχουμε για την ώρα. Και βεβαίω όπω είπα, περιμένουμε και άλλα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν. Όλα αυτά υπόκεινται στον κανονισμό EFSD. Πρέπει να τηρήσουμε τις διαδικασίες που προβλέπει ο κανονισμός. Κάθε δηλαδή συμβολή πρέπει να πάει στο στρατηγικό ε, συμβούλιο που πρέπει να, μετά, αποφασίσει και μετά από τη λήψη την απόφαση εκεί μπορούμε να δεχτούμε τη συμβουλή ή όχι. Εσείς είστε τμήμα, ε, κομμάτι του Στρατηγικού Συμβουλίου και θα βασιστούμε στη δική σας θέση, αλλά πέρα από τον ορισμό και τα άρθρα του κανονισμού, όπου τα κρατη μπορούν να δηλώσουν για συμβολές ανάλογα με τον τομέα ή την περιφέρεια, όπως λέει και ο κανονισμός, θα έλεγα πως οι σύμβολες αυτές δεν φέρνουν μαζί τους οποιαδήποτε προνόμια. Αυτό για τη δική σου ερώτηση. Και τώρα το GTAC είναι κομμάτι της, ε, ε, του κανονισμού, για να απαντήσω σε εσά κύριε Φρουντσουλίκα, είναι το τεχνικό κομμάτι, αλλά η ΕΤΕΠ μπορεί όντω να γνωμοδοτήσει για τα παράθυρα, αλλά όχι για συγκεκριμένα έργα. Ε, Αυτό που μπορούν να κάνουν είναι στο πλαίσιο του GTAC να μας δώσουν την εκτίμηση κινδύνου για τα συγκεκριμένα project για τα μεμονωμένα project. Δυστυχώ, οι διαπραγματεύσει για το GTEC γίνονται εδώ και πάνω από έξι μήνε με την ΕΤΕΠ. Θα θυμάστε ίσω ότι οι σχέσει στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ήταν αρκετά ε, περίπλοκες και θα έλεγα πως εξακολουθούμε να έχουμε κάποια ζητήματάκια αλλά ε, δημόσια ε, εκφράζω την ελπίδα εξ ονόματος της Επιτροπής ότι θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε τελική συμφωνία στα τέλη Απριλίου, δηλαδή μέσα σε αυτή τη εβδομάδα. Και να έχουμε και την αξιολόγηση του κινδύνου από την GTAC μέσα στο Μάιο για να μπορέσουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα που σας είπα στην αρχή της εισήγησής μου. Αλλά είμαι βεβαία και η Κατερίνα έχει να προσθέσει κάτι. Ναι, θέλω μόνο μια διευκρίνηση πριν δώσω το λόγο στην Κατερίνα. Λοιπόν, Είμαι κράτο μέλο λοιπόν. Ξέρω ότι το συζητήσαμε στον τριμερή, αλλά είμαι κράτο μέλο. Έτσι και δίνω ένα εκατομμύριο ευρώ όπω η Γερμανία. Μετά όμω αποφασίζω πού θα πάνε τα χρήματα αυτά. Υπάρχει κάποιο μηχανισμό για να κρίνουμε την προσθετικότητα των κονδυλίων που έρχονται από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Γιατί μπορεί, ας πούμε, η Γερμανία ούτως ή άλλως να πανούσε αυτό το εκατομμύριο. Ενώ αν το περάσει από την Ευρώπη να έχει πιο ευρωπαϊκή εικόνα. Δεν κατηγορώ τη Γερμανία, απλώς παράδειγμα το φέρνω. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία η ευρωπαϊκή Γίνεται πιο συντονισμένα αυτή η συμβολή. Ε, είναι, πιο, είναι κομμάτι ενός ευρωπαϊκού συστήματος. Ο Γκέιτς ε, είναι 42 φορές το ποσό που έδωσε η Γερμανία. Φανταστικό. Και εντάξει, η Γερμανία δίνει με το παραπάνω στον προπολογισμό του, της Ένωσης. Ε, αλλά, εν πάση περιπτώσει, ένα ιδιωτικό ίδρυμα συμβάλλει έχει λόγο για το πού θα πάνε αυτά τα χρήματα. Γιατί αφού το Στρατηγικό Συμβούλιο υπάρχει, τι αποφασίζει αν τα χρήματα αποφασίζει ο δωρητής που θα πάνε. Μπορείτε να μου απαντήσετε αυτό και μετά θα δώσουμε το λόγο και στην κυρία Μεσανόβα. Λοιπόν, να διευκρινίσω. Ακόμη και αν πούνε ότι είναι προκαθορισμένη η χρήση των ε, πόρων πρέπει να πληρούνται όλα τα αντικειμενικά κριτήρια που, που αναφέρει ο κανονισμός. Αυτό ισχύει ακόμη και αν οποιοδήποτε δωρητής κάποιο κράτος μέλος θέλει να προκαθορίσει τη χρήση των πόρων που ε, δίνει. Γιατί αν δεν βασίσουμε την απόφασή μας σε αυτά τα κριτήρια τότε κάτι κάναμε λάθος. γίνεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια. Αν κάποιο κράτος μέλος ούτως ή άλλως ε, χρησιμοποιήσει πόρους ε, που ήδη έχει αποφασιστεί που θα δοθούν, αυτό είναι άλλο. Το συζήτησα όμως πρόσφατα με την EBRD για τη νέα δομή και τη νέα αναπτυξιακή πολιτική μέσω καινοτόμων χρηματοδοτήσεων. Δηλαδή, δεν υπάρχουν επαρκείς δημόσιοι πόροι για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των απεισωμένου κόσμου. Και ξέρετε ποια είναι η εκτίμηση για τους ε, ε, στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Χρειαζόμαστε 3 εκατομμύρια. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξουν και ιδιωτικέ επενδύσεις. Και αυτή είναι η πρώτη φορά που κάνουμε κάτι για να υπάρξει αυτή η προσθετικότητα. Δηλαδή να μοχλεύσουμε ιδιωτικούς πόρους για την ανάπτυξη. Πρέπει λοιπόν να επιτύχει αυτό το πρόγραμμα εξωτερικών επενδύσεων. και να δούμε αν αυτό το μοντέλο μπορεί να είναι η βάση για την καινοτόμο χρηματοδότηση και στο μέλλον. Και νομίζω ότι θα μας βοηθήσουν και τα κράτη-μέλη. Αλλά φυσικά περιμένουν να δουν τα πρώτα αποτελέσματα. Όπως και εσείς. Για να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Ο κύριος Φουντζούλικα. λάβατε προτάσεις από τις χώρες ε, γειτονίας, ιδιαίτερα τις χώρες της ανατολικής συνεργασίας. Γιατί αυτό το μέσο πολλοί νομίζουν ότι είναι μόνο για την Αφρική. Πήγα πρόσφατα στο Κίσινο και στο Κίεβο. Πριν από δύο εβδομάδες. Οι αρχές εκεί δεν έχουν ιδέα για αυτό το μέσο. Μήπως πρέπει να τους το γνωστοποιήσετε. Σωστό, ωραία. Η Digineer να απαντήσει. Ευχαριστώ. Πολύ καλή ερώτηση είναι αυτή. Το Κίσινάου περιμένουμε ακόμη να μας στείλει κάποιες προτάσεις, αλλά οι αρχές και των έξι χωρών της Ανατολικής Γειτονίας έχουν ενημερωθεί επανειλημμένα, έχουμε συζητήσει επανειλημμένα και μέσω διπλωματικών διάβλων, αλλά και προσωπικά πήγα και στο Κίεβο και στην Τυφλίδα για να παρουσιάσω το πρόγραμμα αυτό στις χώρες και θα πάω και στο Κίσινα προσεχώς μόλις ε, επιληθεί η πολιτική κρίση θα συνεχιστεί η διαδικασία και με το Ερεβάν Είμαστε σε επαφή και με την κυβέρνηση του Μπελαρούς. Και αυτή τη βδομάδα ή την επόμενη θα τους παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας κατά τη συνεδρίαση μιας ε, υψηλού επίπεδου ομάδας συντονισμού. Είναι το υψηλότερο επίπεδο συνεργασίας. Βεβαίως μπορεί κάποιες παρουσιάσεις να είπαν ότι κυρίως αφορά την Αφρική αλλά έχουμε επανειλημμένα υπενθυμίσει τους εταίρους μας της Ανατολικής Γειτονίας ότι βεβαίως καλύπτει και την περιοχή τους και τον Νότο. Πολλές προτάσεις από τους εταίρους μας αφορούν χώρες γειτονίας. Έχουμε τρεις είδους προτάσεις για τα PIPS που ανέφερε η Μαριέτα. Ορισμένες είναι μόνο για την Αφρική, ορισμένες είναι μικτές και ορισμένες είναι αποκλειστικά για τη γειτονία. Καλύπτουμε δηλαδή πλήρως. Με συγχωρείτε που ήρθα με καθυστέρηση λίγο λεπτό υποθέτω ότι η Μαριέτα θα ανέφερε ότι για τις προτάσεις ε, για τα δύο πρώτα, τις δύο πρώτες χρηματοδοτήσεις έχουμε ήδη υπερκαλύψει. Και για τις τρεις επόμενες χρηματοδοτήσεις, τα τρία επόμενα παράθυρα χρηματοδοτήσεων, όπως θα λέμε, ήδη έχουμε καλύψει τα ποσά μέσω των προτάσεων. Άρα θα έχουμε μερικές ε, έντονες συζητήσεις με τους εταίρους μας για να τους πείσουμε να συνεργαστούν και να κάνουν και πιο ε, λελογισμένες προτάσεις για κάποιες εγγύησεις. Τώρα, Κάποιες ερωτήσεις που ετέθησαν προηγουμένως. Σύμφωνα με τον κανονισμό, τα κράτη-μέλη, όχι οι ιδιωτικοί συνεργαζόμενοι, τα κράτη-μέλη μπορούν να κάνουν στόχευση και ε, θεματική και γεωγραφική. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει, γιατί τα ποσά είναι κάπως συμβολικά, αλλά επειδή είναι μικρά τα ποσά, εύκολο είναι να τα, ε, να τα ορίσουμε για κάποιο συγκεκριμένο στόχο, να μην υπάρξει μεγάλος ε, κατακαιρματισμός. Εάν κάποιο κράτος μέλος ε, συμβάλλει περισσότερο, θα δούμε πώς θα αποδοθούν οι χρηματοδοτήσεις. Λοιπόν, πρέπει να τελειώσουμε 6,5 ακριβώς ο κύριος Αρτουή και μετά ο Ζων Χάουζ. Ευχαριστώ. Θέλω λίγο περισσότερα για τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που υποτίθεται ότι θα συνέβαλε με την τεχνογνωσία της. Τι γίνεται. Γιατί η καινοτομία είναι ότι μπορεί οποιοδήποτε θέλει να χρηματοδοτήσει μπορεί να χρηματοδοτήσει ε, ενοχλήθηκε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δημιούργησε προβλήματα. Λέμε επίσης ότι Α, λέμε ότι οι μεγάλες εταιρείες Google, Apple και τα λοιπά, Facebook θα πρέπει να πληρώσουν περισσότερο γιατί δεν πληρώνουν αρκετούς φόρους στην Ευρώπη. Η Εστονία, η Τσεχία και η Γερμανία επίσης συμβάλλουν. ενώ δεν συμβάλλουν για να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για το χρηματοδοτικό μέσο για την Τουρκία. Η χρηματοδοτική διευκόλυνση. Είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Παίρνουμε λεφτά από την Τουρκία και τα δίνουμε για αυτό το νέο μέσο. Δεν θα ήταν πιο απλό το σύνολο των κρατών για μια φορά να συμφωνήσουν. Τα θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι τεράστια και για την μετανάστευση δεν ξέρουμε ακόμη τι θα μας έρθει στο κεφάλι. Θα πρέπει να καταλάβουν τα κράτη-μέλη τι δεσμεύσει πρέπει να αναλάβουν για τα θέματα αυτά. Και μία ερώτηση. Οι κομόρες συμμετέχουν στο, στο πρόγραμμα γιατί η μετανάστευση από τις κομόρες στο... στην Ίσο Μαγιότ είναι σημαντική. Ευχαριστώ. η Επιτροπή μας έκανε κατανομή κατά κλάδο. Μήπως έχουμε μια παρόμοια γεωγραφική κατανομή. Λοιπόν, ένα σχόλιο ακόμη. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερους πόρους για την ανάπτυξη. Αλλά εξήχθησαν διδάγματα από τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη χώρα μου επειδή υπάρχει μεγάλη ανάγκη για νέα νοσοκομεία και νέα σχολεία, πριν από 15 χρόνια επιτρέψαμε πολλές μικτές χρηματοδοτήσεις. Λεγόντουσαν PFI. Ο ιδιωτικό τομέα εκτίζει ένα σχολείο και ένα νοσοκομείο και μετά το δανείζει στο δημόσιο. Αλλά τι έχει συμβεί. Τα δάνεια αυτά τα πουλάνε και τα ξαναπουλάνε, έχουν γίνει πολύ ακριβά και το κόστος τώρα για το δημόσιο κορβανά είναι πολύ ψηλότερο από ότι θα ήταν εάν το κράτος είχε δανειστεί αυτά τα λεφτά για να χτίσει το σχολείο. Τα έχει δανειστεί στην αγορά, θα ήταν πολύ φθηνότερο. Εξήχθησαν λοιπόν διδάγματα από τα λάθη του παρελθόντος και έχουν ουσιώδεις επιπτώσεις. Τα σχολεία στην πόλη μου που χτίστηκαν με αυτό το σύστημα θέλουν να χτίσουν ε, μία νέα αίθουσα, κυνηγάνε τραπεζίτες στην Ελβετία και στη Γαλλία για να χτίσουν μια νέα αίθουσα διδασκαλία στο Σέφιλ. Να μην ξανακάνουν τέτοια λάθη. Ελπίζω να έχει μάθει κομισιόν. Δεν υπάρχει δωρεάν χρήμα. Το χρήμα πάντα κοστίζει και κάποια στιγμή θα το πληρώσει. Δεν ξέρω πώ να απαντήσει σε Μαριέτα, θα επιχειρήσω. Έχουμε έξι λεπτά. Σχέση με την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Όπως σε κάθε οικογένεια οι σχέσεις είναι περίπλοκες, αλλά φυσικά πολύ καλές. Έχουμε καθημερινή συνεργασία. Και υπάρχουν κάποια προβληματάκια. Αλλά για το GTEC λοιπόν έχουμε προβλήματα όπου έχουμε κάνει την αναγκαία συμβατική εργασία με όλους τους άλλους θεσμούς. Η ΕΤΕ λοιπόν θα χρηματοδοτήσει μερικά καινοτόμα BIPs που θα αξιολογηθούν με τα ίδια κριτήρια. Όπως όλα τα BIPs και θα γίνει αυτή η εξέταση, όπως είπα, μαζί με τα άλλα BIPs. Για τη γραφική κατανομή δεν μπορώ να σας δώσω την ίδια κατανομή όπως τη θεματική κατανομή γιατί εκτός από τις γειτονικές χώρες Αφρικής τα BIPs αναφέρονται σε συγκεκριμένη περιφέρεια λένε είτε η Αφρική ή η γειτονία θα θέσουμε περαιτέρω ερωτήσεις στις ε, προπαρασκευαστικές ερωτήσεις που θέλετε να χρηματοδοτήσετε κάτι τι προστατικότητα θα υπάρχει. Και όταν το κάνουμε αυτό, τότε νομίζω ότι θα σας δώσουμε και αυτή τη γεωγραφική κατανομή. Για τις Κομόρες, ναι βεβαίως, ανήκουν στο Κοτονού, άρα είναι επιλέξιμα. Αυτά. Το ιδιωτικό τομέα ξέρουμε τους κινδύνους της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα αλλά θεωρώ ότι η μόχλευση πρέπει να είναι σωστά προσανατολισμένη ούτω ώστε οι τελικές αποφάσεις τελικά να παίρνονται από τους θεσμούς που είναι υπόλογε στον Ευρωπαίο πολίτη. Ευχαριστώ. Κυρία Μαρτένο, έχετε να προσθέσετε. Πολύ καλά τα σχόλια του κυρίου Αρτουή. Βεβαίως θέλουμε να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη για να μην παίρνουμε από τον έναν για να δώσουμε στον άλλον. Και αυτό βεβαίως είναι μια πρόκληση για όλους μας. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Α, εντάξει, πήρα την απάντησή σας. 18-27, κερδίζουμε και 3 λεπτά. Ωραία, ολοκληρώνω τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ την Επιτροπή για την παρουσία της. Το θέμα αυτό θα το παρακολουθήσουμε και περαιτέρω. Ευχαριστώ πολύ.